Witam bardzo serdecznie. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι γιατί μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που ε, θέμα έχει την προφορική ερώτηση για την θανατική ποινή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην συντάκτρια της ερώτησης αυτής, την κυρία Ελένα Βαλενσιάνο. Παρακαλώ. Gracias, Στις 10 του μηνός είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ανητικής ποινής και είναι